Η διάταξη είναι η παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και η δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Συμβούλιο Κορυφής της 29ης και 30ης Οκτωβρίου σχετικά με την εντολή και τις αρμοδιότητες του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου όπως επίσης και του υπάτου εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και την πολιτική της ασφάλειας όπως επίσης και για τη διάθρωση της νέας Επιτροπής. Είμαι ευγνώμων λοιπόν προς τον Πρωθυπουργό κ. Ρέινφελτ και τον Πρόεδρο κ. Μπαρόσο. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Πρωθυπουργό. Κύριε Φρέντρικ Ράινφελτ, έρχεται το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη, με μεγάλη χαρά είμαι ανάμεσά σας σήμερα. Θα ήθελα να σας μεταφέρω το τι συνέβη σε ένα περίπλοκο θα έλεγα συμβούλιο. Να ξεκινήσω λέγοντας τι έγινε λίγο πριν από τη συνεδρίαση. Ήμασταν σε μόνιμη επαφή με την Πράγα, πώς θα λύναμε το πρόβλημα και το αίτημα των Τσέχων σχετικά με τη χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Υπήρχαν διαφορετικές απόψεις και αιτήσει για πολλές ε, ε, εξαιρέσεις Αντίθετα είχαμε ένα πιο ξεκάθαρο μήνυμα για τις κλιματολογικές αλλαγές. κρατημέλη δεν ήταν έτοιμα να καταλήξουν σε συγκεκριμένα ποσά για την χρηματοδότηση μέσων προσαρμογής και αντιμετώπισης των συνεπειών στις αναπτυσσόμενες χώρες. Παρ' όλα αυτά λοιπόν και λόγω όλων αυτών των θεμάτων είμαι γενικά ικανοποιημένος από το πώς πήγε η συνάντηση αυτή. Στόχος μας, μιας και πλησιάζουμε στη συνάντηση της Κοπενχάγης για το κλίμα, έπρεπε να συζητήσουμε ορισμένα θέματα. Οι διαπραγματεύσεις ήταν δύσκολες, οι διαπραγματεύσεις κράτησαν αρκετά, αλλά στο τέλος υπήρξε έγκριση από πλευράς του Συμβουλίου της πρόβλεψης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 100 δις κατέτος μέχρι το 2020 θεωρείτε ότι η διεθνής συνεισφορά θα πρέπει να φτάσει στο συγκεκριμένο έτος από 22 με 50 δις. Βέβαια το 2020 δεν είναι και πάρα πολύ μακριά και πέραν τούτου θα υπάρξει και συνολική χρηματοδότηση 5 με 7 δις κάθε χρόνο από το 2010 μέχρι το 2012. Ένα τελικό ποσό για το κόστος αυτής της παρέμβασης ε, θα καθοριστεί στα πλαίσια της συνάντησης της Κοπενχαΐς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να κάνει τη δική της συνεισφορά εφόσον και άλλοι ε, βασικοί παίκτες στη διεθνή σκηνή κάνουν αντίστοιχες προσπάθειες. Εδώ και λίγες μέρες Επέστρεψα μετά από διαπραγματεύσεις ε, με τον Πρωθυπουργό Σίνγκ στη συνάντηση κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Ινδίας στο Νέο Δελχή. Και την προηγούμενη εβδομάδα είχα επαφές ε, με τον πρόεδρο Ομπάμα στη συνάντηση κορυφής ε, στη Ουάσιγκτον. Ακριβώς χάρη στη συμφωνία της σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν σε θέση να διαπραγματευτεί τα θέματα αυτά με πολύ συγκεκριμένη άποψη. Παρουσιάσαμε αξιόπιστα τις απόψεις μας, μπορέσαμε να ενθαρρύνουμε τους συνομιλητές μας και για μια ακόμη φορά είμαστε ικανοί να καθοδηγήσουμε τη συζήτηση αυτή, ένα θέμα κρίσιμο για όλους τους πολίτες. Το θέμα αφορούσε βέβαια και την οικονομική και χρηματοπιστωτική κατάσταση. Βέβαια υπάρχουν δείγματα, ενδείξεις μάλλον, βελτίωσης της παγκόσμιας οικονομίας, αλλά δεν υπάρχει προς στιγμή τουλάχιστον χώρος για καθησυχασμό. Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός από μία ίσως, θα ξεπεράσουν το 3% του ανωτάτου ορίου για το έλλειμμα. Αυτοί είναι λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να συνεχιστούν τα μέτρα τα οποία έχουμε λάβει για την αντιμετώπιση της κρίσης. Και θα προσπαθήσουμε εν τω μεταξύ να επεξεργαζόμεθα και τις στρατηγικές εξόδου από την κρίση. Κάναμε βήματα πρόοδου και στα πλαίσια της ενίσχυσης της ε, επίβλεψης των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών όπως επίσης συζητήσαμε και την δημιουργία της Επιτροπής ή της Ομάδας Αξιολόγησης Συστημικών Κινδύνων ή Συστημικού Κινδύνου. Θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε μια νέα χρηματοπιστωτική κρίση σαν αυτήν την οποία βιώνουμε τώρα. Όταν όλα ξεκινήσουν να λειτουργούν, βασικό μα στόχο θα πρέπει να είναι η διατήρηση των θέσεων απασχόληση. Άνω των 5 εκατομμυρίων Ευρωπαίων έχασα τι θέσει του και πολλοί από αυτού αντιμετωπίζουν την προοπτική τη ανεργία. Πρέπει να ανταλλάξουμε όλα αυτά. Παρουσίασα τι προτεραιότητε τη Σουηδικής Προεδρία στι 15 Ιουλίου και είπα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βγει ενισχυμένη από την κρίση αυτή και ακριβώ βασική πρόκληση για μα ήταν η διαχείριση τη οικονομική κρίση και εξακολουθεί να είναι. Γι' αυτό τον λόγο λοιπόν θα επανέλθουμε σε αυτά τα σημαντικά θέματα στη συνάντηση κορυφή τον μήνα Δεκέμβριο. Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, ένα πολύ σημαντικό θέμα που συζητήθηκε επίση ήταν η υιοθέτηση τη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την περιοχή της Βαλτική θάλασσας. Μια στρατηγική που βασίζεται σε μια πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Φιλοδοξία μας είναι με τη στρατηγική αυτή να αντιμετωπίσουμε τα περιβαλλοντικά προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν στην περιοχή αυτή και να βοηθήσουμε και την οικονομική της ανάκαμψη. Είμαι πεπισμένος ότι η πρωτοβουλία αυτή θα λειτουργήσει θετικά και για άλλα μέρη της Ευρώπης και θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της. Συζητήσαμε επίσης και τα θέματα εσωτερικών υποθέσεων και δικαιοσύνης, Υπήρξαν πρόοδοι σε θέματα όπως η παράνομη μετανάστευση στην Μεσόγειο και ζητήσαμε να γίνουν περαιτέρω έρευνες και προσπάθειες σε συγκεκριμένους τομείς. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, υπάρχουν θέματα θεσμικά, συνταγματικά που θα θέλατε να συζητήσετε σήμερα το απόγευμα και αυτά ήταν ένα από τα θέματα που συζητήσαμε. Συζητήσαμε τον τρόπο έτσι ώστε να τεθεί σε ισχύ το ταχύτερο δυνατόν η συνθήκη της Λισαβόνας. Αυτό είναι κρίσιμο για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας μαζί. Οι διαπραγματεύσεις ήταν ε, σε αρκετά επίπεδα και ήταν αρκετά περίπλοκες. Στο τέλος καταφέραμε να δεχθούμε τα αιτήματα της τσεχικής δημοκρατίας και ο πρόεδρος Βάκλαβ Κλάους ήταν προετοιμασμένος να υπογράψει την συνθήκη και όπως όλοι γνωρίζετε το έκανε εδώ και μία εβδομάδα. Το τελικό μέσο λοιπόν της επικύρωσης έχει ήδη κατατεθεί και από την τσεχική ε, δημοκρατία στις Ιταλικές αρχές. Αυτό σημαίνει ότι η συνθήκη της Λισαβόνας θα τεθεί σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου. Γνωρίζω ότι η μεγάλη πλειοψηφία από όλους τους παρόντες εδώ σήμερα συμμερίζεται την δική μου ικανοποίηση και ανακούφιση αν θέλετε αυτό το προπαρασκευαστικό κεφάλαιο έχει αρχίσει να ολοκληρώνεται πλέον. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αξιολόγησε επίσης και άλλα προπαρασκευαστικά βήματα για τη συνθήκη, συμφώνησε στις κατευθυντήριες γραμμές για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, και ζήτησε και θα ζητήσει από τον μελλοντικό ύπατο να παρουσιάσει προτάσεις για την οργάνωση της υπηρεσίας αυτής. Τώρα να έρθω στα ονόματα. Πρέπει να έχουμε ε, διορίσει τους συγκεκριμένους, ε, τον πρόεδρο δηλαδή και την Επιτροπή και τον ύπατο πάρα πολύ σύντομα. Στις 19 ε, Νοεμβρίου θα γίνει μια συνάντηση αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων έτσι ώστε να καταλήξουμε στον κατάλογο των ονομάτων. Ο διορισμός του υπάτου εκπροσώπου θα πρέπει να γίνει πριν από το διορισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αυτό θα πρέπει ε, να γίνει επίσης μετά από επαφές και με το κοινοβούλιο σας. Το συγκεκριμένο πρόσωπο θα είναι έτσι κι αλλιώ και αντιπρόεδρο τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γι' αυτό αυτό ή αυτή θα πρέπει να εγκριθεί και από το ίδιο κοινοβούλιο μετά από ψηφοφορία του. Δεν θα περάσω τώρα στο να λέω ποια μπορεί να είναι τα συγκεκριμένα ονόματα. Αλλά το θέμα δεν είναι το όνομα. Το θέμα είναι το τι θα κάνουν οι συγκεκριμένοι αυτοί οι πολίτες και πώς θα το κάνουν. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λοιπόν της προηγούμενης εβδομάδας μας βοήθησε να προχωρήσουμε όχι μόνο σε ένα αλλά σε πολλά θέματα. Θέματα τα οποία είναι ζωτικά για το μέλλον της Ευρώπης, ζωτικά για το μέλλον του πλανήτη. Είμαι ευγνώμων προς τους συναδέλφους μου για την επικοδομητική του στάση απέναντι στις προκλήσεις που από κοινού αντιμετωπίζουμε. Βέβαια γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε. Σας υπόσχομαι ότι τις επόμενες εβδομάδες θα είμαστε όλοι ιδιαιτέρως απασχολημένοι. Θα συνεχίσω την συνεργασία μου με το Κοινοβούλιο, την στενή συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Η συνάντηση στην Κοπενχάγη ξεκινάει μόνο σε, σε 25 μάλλον μέρες και η οικονομική κρίση δεν έχει ακόμα τερματιστεί. Παρ' όλα αυτά έχουμε πλέον μια σαφέστατη εντολή στις διαπραγματεύσεις για το κλίμα. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεργαστούμε, να οδηγήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση σε υψηλότερα επίπεδα απασχόλησης και ε, φυσικά εδώ μετράω και τη δική σας υποστήριξη. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Prime Minister. Σας ευχαριστούμε, κύριε Πρωθυπουργέ. Καλώ τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο, στο βήμα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Θα ήθελα να συγχαρώ τον Πρωθυπουργό Ράινφελ για την αξιολόγηση που έκανε για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Σχολίασε την, ε, τα θέματα πολιτικής και τα θεσμικά θέματα. Το βασικό αποτέλεσμα που όλοι περιμέναμε για την πολιτική ήταν η απόφαση για την ε, πολιτική καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Πολλά διακυβεύονται και σίγουρα θα είναι δύσκολος ο δρόμος. Αλλά πραγματικά υπερεύει τις αρχικές προσδοκίες μου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τελικά εγκρίθηκαν τα ποσά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με μια ισχυρή αιρεσιμότητα. Και είναι σαφές ε, το μήνυμα, είμαστε έτοιμοι για την Κοπενχάγη έτοιμοι για να μειωθούν οι εκπομπές και να χρηματοδοτήσουμε αυτές τις προσπάθειες όπως πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Σεπτέμβριο και μακρό πρόθεσμα και ευραχή πρόθεσμα. Γιατί αν οι αναπτυσσόμενε χώρε θέλουμε να έρθουν στο των διαπραγματεύσεων με ισχυρέ δεσμεύσει για άμβλυνση των κλιματικών αλλαγών, θα πρέπει να κάνουμε και εμεί σοβαρέ προτάσει από πλευρά ανεπτυγμένων χωρών. Μέχρι το 2020 θα χρειάζονται 100 δι ευρώ για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών το χρόνο και αυτό υποστηρίχθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Υπάρχει γενικότερη υποστήριξη από την διεθνή κοινότητα και ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικά θα υποβάλει την δέουσα εισφορά. Και οι άλλοι εταίροι πρέπει να καταδείξουν ε, ότι παίρνουν στα σοβαρά τις προθέσεις μας. Η πολιτική μας ε, δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να χαράξει το δρόμο ελπίζοντας ότι θα ακολουθήσουν οι άλλοι. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη δύναμη μόχλευσης που έχουμε για να προάγουμε τις διεθνείς προσπάθειες για την μείωση των εκπομπών. Όταν στο Νέο Δελχή την περασμένη εβδομάδα μου υπενθύμησαν ναι, σε ποιο βαθμό έχουν προχωρήσει τον τελευταίο χρόνο οι δύο εταιρείε στον τομέα αυτό. Αυτό ισχύει και για άλλους εταιρείε, όπως ε, για την Κίνα. Φυσικά συνεχίζουμε να τηρούμε τη βασική απέτηση τη ε, διαφοροποιημένη, αλλά κοινή ευθύνη για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Σας έχω πει επανειλημμένα ότι πρόκειται για κοινή προσπάθεια και εμεί ε, ω Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσουμε να πιέζουμε ούτω ώστε όλοι οι υπόλοιποι παίκτε να συνεισφέρουν στη διαδικασία και πρέπει να εστιάσουμε στο στόχο μας. Ε, πρέπει να έχουμε αξιόπιστες, μεγάλε μεγάλες μειώσεις, εκπομπέ, ούτως ώστε να περιορίσουμε την αύξηση της θερμοκρασίας σε λιγότερο από 2 βαθμούς Κελσίου, όπως έχουμε υποσχεθεί. Τι γίνεται εν ώψη της Κοπενχάγης τώρα. Κατά πάσα πιθανότητα δεν θα υπάρξει πλήρη συμφωνία, θα συνεχίσουμε όμως να πιέζουμε και δεν είναι λόγος αυτό για να ε, δεχτούμε οποιαδήποτε υποχώρηση. Μπορεί ε, στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων να γίνουν αποφασιστικά βήματα. Τη σημασία έχει τι θα γίνει στην Κοπενχάγη. Πρέπει να πιέσουμε για τη συμφωνία βασιζόμενη σε ισχυρή πολιτική δέσμευση. Θέλουμε ταχεία θέση σε εφαρμογή τη συμφωνία με συμμετοχή όλων και για τη μείωση των εκπομπών των ρήπων και για τη χρηματοδότηση. Και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την τελική συμφωνία, για μια δεσμευτική συνθήκη. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να συσπηρωθούμε μέχρι, μέχρι να διεξαχθεί η Σύνοδο Κοπενχάγη αξιότιμη βουλευτή Ευρωβουλευτέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μόλι καταδείξαμε ότι με κοινή αποφασιστική δράση μπορούμε να συμφωνήσουμε για μια συνθήκη που θεωρούσαμε ότι δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί. Ε, και αυτό είναι βασική πρόοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Κατέληξε τον τελευταίο φραγμό για την ε, τελική επικύρωση τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Και τώρα μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη γιατί όπως είπε ο Πρωθυπουργό ε, Ράινφελντ θα αρχίσει ε, στη, την 1η Δεκεμβρίου να ισχύει η συνθήκη της Λισαβόνας. Εμείς εργαζόμαστε ήδη για την εφαρμογή της συνθήκης. Αρχίσαμε σήμερα τη διαβούλευση για την πρωτοβουλία των πολιτών. Να, ένα πρώτο απτό βήμα. Από τι οφόρο τιμή στον Πρωθυπουργό Ράινφελτ ε, για την συμμετοχή του στην πρόοδο που σημειώθηκε. Ε, εργαστήκατε με πολύ αξιόλογο τρόπο και συνεισφέρατε στο να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αλλά το θέμα είναι η μετάβαση στη νέα περίοδο. Για τις νέες θέσεις, ε, δεν θα ήθελα τώρα να σχολιάσω εγώ το θέμα των υποψηφίων για τις δύο θέσεις, αλλά με την ιδιότητα του Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για τα θεσμικά ζητήματα, ελπίζω ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα επιλέξουν την προσωπικότητα που μπορεί με αποτελεσματικότητα να ηγηθεί του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα έχει ισχυρή ευρωπαϊκή δέσμευση που θα υποστηρίξει τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού ε, Συμβουλίου με ένα τρόπο. Θα μπορέσουμε έτσι μακροπρόθεσμα να θέτουμε πρωτοβουλίες όχι μόνο ε, για, το επόμενο εξάμεινο και σε εξωτερικό επίπεδο. Η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας ε, θα μπορέσει να περάσει ισχυρά μηνύματα στους εταίρους μας. Ε, και θα συνεργαστούμε με, στενά με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου γιατί αυτό θα κάνει τη διαφορά η καλή συνεργασία. Σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων πρέπει να συστήσουμε μια ΚΕΠΑ όπου ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση στο δικό του επίπεδο και θα πρέπει επίσης ε, να ε, συσπυρώσουμε όλες τις αρμοδιότητες που έχει η κοινότητα στο εμπόριο, στην οικονομία, στη διεύρυνση, για τα ενεργειακά ζητήματα για τα θέματα δικαιοσύνη, ε, για τα οποία σύμφωνα με τη συνθήκη εκπροσωπεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Ένωση ε, θα πρέπει να ε, προάγουμε τις προσπάθειές μας σε ιστορικό επίπεδο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Τώρα θα ήθελα να αναφερθώ στο ότι το πρόεδρος του, ο ύπατος εκπρόσωπος ε, θα είναι επίσης ε, αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο διορισμός του υπάτου εκπροσώπου και οι λοιπές προτάσεις ε, που θα γίνουν για τα υπόλοιπα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα μου επιτρέψουν να καταλήξουμε σε απόφαση στην επόμενη σύσκεψη του σώματος και ο αντιπρόεδρος ε, ε, θα ε, υποστηρίζει, θα επικουρείται από μια ισχυρή υπηρεσία για την εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε στα διπλωματικά θέματα και με την αρμοδιότητα που έχουμε να φέρουμε την αλλαγή ως προς την εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να απαρτίζεται από αφοσιωμένους Ευρωπαίους με τα κατάλληλα προσόντα για να εξασκήσει το δικαίωμα πρωτοβουλία που έχει και στι τελευταίε συζητήσει που έχω με τα κράτη-μέλη με ρημνό, ώστε να ισχύσουν αυτά. Θέλω να μου προτείνουν άντρε και γυναίκε ε, τα κράτη-μέλη για υποψηφίου και υποψήφιε ε, για να ε, τα χαρτοφυλάκια, για τα χαρτοφυλάκια ανήκουν σε αυτά τα άτομα και όχι στα κράτη-μέλη, σε αυτά τα άτομα που έχουν αυτή την ισχυρή δέσμευση. Οι καθυστερήσεις που έχουν σημειωθεί λόγω της συνθήκης συνιστούν κοινή πρόκληση. Δεν πρέπει να καθυστερήσουμε πλέον, θέλουμε σύντομα την νέα επιτροπή, αλλά δεν μπορούμε να παρακάμψουμε και τις ακροάσεις που πρέπει να διεξαχθούν. Αυτό θα συζητηθεί την ερχόμενη εβδομάδα στη διάσκεψη των Προέδρων. Χάρη συνθήκη συνθήκες Λισαβόνας μπορούμε να καλύψουμε περισσότερο τις προσδοκίες των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά πάνω απ' όλα, όλα είναι ζήτημα πολιτικής θέλησης και η συνθήκη Μα δίνει το δικαίωμα να ενεργήσουμε. Αλλά πριν ενεργήσουμε θέλουμε και κοινή πολιτική βούληση για κοινή δράση ε, η Ευρώπη όπως εκπροσωπείται εδώ σήμερα είναι μια ενωμένη Ευρώπη με ελευθερία και αλληλεγγύη. Αυτό δεν θα ήταν δυνατό χωρίς την αφοσίωση και τη δέσμευση αυτών που έκαναν ε, ε, καταπληκτικά επιτεύγματα στις απαρχές Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και ε, αν σήμερα το 2009 δείξουμε την ίδια αφοσίωση σίγουρα θα επιτύχουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε της Κομισιόν. Τώρα θα λάβουν το λόγο οι εκπρόσωποι από τις πολιτικές ομάδες. Καταρχήν από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και Ευρωπαίοι ο κύριος Ντόλ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, έχει κυρωθεί η συνδίκη της Λισαβόνας από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρώπης και τώρα είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε και να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Όλα αυτά εξαρτώνται από την ταχεία κάλυψη των θέσεων ευθύνη. Είμαστε υποχρεωμένοι επίση να έχουμε θετικά αποτελέσματα για το κλίμα και την ενέργεια. Επίση και κυρίω για την οικονομική ανάκαμψη. Με την υπογραφή του Βάτσλαβ Κλάου, η διαδικασία κύρωση τη συνθήκη συνθήκης Λισαβόνας επιτέλους τελείωσε και πέρα το είχε χάρη στον Φρέντερικ Χάινφελ. Η ομάδα του ΕΛΚ, η οποία έχει σφραγίσει με την παρουσία της τη συνθήκη τη Λισαβόνα, είναι ικανοποιημένη. Αλλά δεν θέλουμε πια να συνεχίσει η δημόσια συζήτηση στην Ευρώπη να στρέφεται μόνο γύρω από του θεσμού τη Ευρώπη και θα πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μα στις πραγματικέ φιλοδοξίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό, κύριε Ράινφερντ, εμεί θέλουμε να επιτύχουμε μια συμφωνία το ταχύτερο δυνατό για το όνομα του Προέδρου του Συμβουλίου και του Προέδρου και του ΙΠΑ του εκπροσώπου. Γι' αυτό ζητάει η ομάδα μου, κύριε Μπαρόσο, από εσύ που τα κράτη-μέλη θα έχουν καθορίσει του υποψηφίου του, να υπάρξει η ταχύτερη δυνατή κατανομή των χαρτοφυλακίων πριν γίνει η διαδικασία ακρόαση των υποψηφίων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που θέλουμε να είναι μια πλήρη ακρόασή του. Προφανώ, κύριε Πρόεδρε, του Συμβουλίου και κύριε Πρόεδρε της Κομισιόν γνωρίζετε ότι το θέμα των επιτρόπων δεν ενδιαφέρει μονάχα το μικρό κόσμο των Βρυξελών αλλά 500 εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών. Τι θέλουν οι πολίτες μας. Θέλουν να αντιμετωπιστεί η ανεργία, να υπάρχουν πιστώσεις, να υπάρχει καλύτερη κατάρτιση, να υπάρχουν αποτελέσματα στην Κοπενχάγη, να μπορέσουμε <clears throat> να μην υπάρχει και πάλι διακοπή εφοδιασμού σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο στην, το χειμώνα του 2009 που θα οδηγήσει σε μεγάλα προβλήματα την Ήπειρό μας. Βρισκόμαστε σε μια κομβική στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Ράινφελτ, όπως τονίσατε και εσείς, πρέπει να κινηθούμε με ταχύτητα τρένου υψηλή ταχύτητα και όχι με ταχύτητα καρβουνιάρα. Όλοι ξέρουν πόσο μεγάλε είναι οι δυσκολίε για να μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτή την ισορροπία μεταξύ των πολιτικών απόψεων, των εθνικών ευαισθησιών και επίσης τη διαθεσιμότητα προσωπικότητων. Αλλά πρέπει και είναι καθήκον σα εσείς να επιτύχετε το ταχύτερο μια συμφωνία στο Συμβούλιο, όπως είναι και καθήκον του Κοινοβουλίου και των πολιτικών ομάδων να μπορέσουν να εκφέρουν άποψη για τις επιλογές αυτές με ένα υπεύθυνο τρόπο και με σεβασμό του γενικού ευρωπαϊκού συμφέροντος. Ελπίζω ότι θα μπορέσει να γίνει πραγματικότητα μέσα στη Σουηδική Προεδρία και να είναι ένα από τα επιτεύγματά τη. Για να γίνει κάτι τέτοιο όμω πρέπει να δράσετε πολύ ταχαίω κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πολύ περισσότερο από τους θεσμικούς όρους αυτή τη στιγμή πιέζει την Ευρωπαϊκή Ένωση το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Βρισκόμαστε πολύ κοντά στη συνδιάσκεψη της Κοπεχάγης. Θέλω να χαιρετήσω το θετικό πνεύμα του ε, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που τονίζοντας τη δέσμευσή της για τη μείωση της εκπομπής διοξιδίου του άνθρακος και της ε, κλιματικής αλλαγής περιμένει την ίδια αποφασιστικότητα και δέσμευση και από τους εταίρους μας. Θα ήταν λαθασμένη τακτική για την Ευρώπη να κατεβάσει όλους τους φραγμούς και να ανοίξει τα χαρτιά της, ενώ οι Αμερικανοί, οι Κινέζοι, οι Ινδοί και οι άλλες χώρες δεν λαμβάνουν υπόψη καθόλου αυτή την υποχρέωση. Οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Κίνα και η Ινδία σαν παγκόσμιες δυνάμεις πρέπει να αναλάβουν και αυτές τις ευθύνες τους όπως τις υπομίζεται η Ευρώπη, η οποία όμως δεν μπορεί να λύσει μόνη στα προβλήματα του πλανήτη. Στην Κοπενχάγη δεν αρκεί μια πολιτική συμφωνία, χρειάζεται να υπάρξει πραγματική δέσμευση και συγκεκριμένη σε ποσοτικό επίπεδο όλων των κρατών μερών. Και σας λέω αγαπητοί συνάδελφοι, είμαστε υποχρεωμένοι να πετύχουμε. Αυτή η υποχρέωση αφορά πρώτα απ' όλα την οικονομική ανάκαμψη και την απασχόληση γιατί είναι αλληλένδετα αυτά τα δύο. Ακόμα και αν φαίνεται ότι αρχίζει πάλι μια μικρή ανάκαμψη, είναι απαραίτητο να δούμε ότι αυτή η ανάκαμψη θα συνοδεύεται με τη δημιουργία θέσεων απασχόληση και αν και θα είναι απαραίτητο επίση να βασίζεται σε υγιή, σε υγιείς βάσεις, σε μια αγορά η οποία είναι ανοιχτή, ρυθμιζόμενη και όχι προστατευτική. Αυτό είναι που ενδιαφέρει τους, Ευρώ, τους Ευρωπαίους, αυτό πρέπει να ενδιαφέρει την Ευρώπη και τα κράτη-μέλη και όχι μονάχα τα θέματα των προσώπων και της εμμελητίας. Γιορτάζουμε τα 20 χρόνια της ε, πτώσης του τείχους του Βερολίνου ήταν η ανθρώπινη θέληση που οδήγησε σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Είναι λοιπόν η στιγμή, κύριε Ράινφελτ, να πείσετε τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε του ΕΛΚ, τώρα εξ ονόματος της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Έχει το λόγο ο κύριος Χάνης Βόμποντα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Κομισιόν. Ίσως είναι μια ευτυχή συγκυρία ότι η συζήτηση αυτή στην οποία ήταν παρόν και ο Βάτσλαβ Χάβελ λαμβάνει υπόψη αυτή τη στιγμή που είναι τόσο σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να γνωρίζει την σημασία αυτής της στιγμής για το μέλλον της. Εγώ γεννήθηκα 20 χιλιόμετρα μονάχα από τα σύνορα στην ε, σε μία από τις δυτικές ζώνες ε, κατοχής τότε, πολύ κοντά όμως στα σύνορα. Και βλέπω ότι η συνδίκη της Λισαβόνας είναι μια πραγματική νέα διάσταση σε αυτή τη διαδικασία που οδήγησε στη σημερινή Ευρώπη. Ήταν απαραίτητο να υπάρξει βέβαια αυτή η υπογραφή του Βάτσλαφ Κλάους και ίσως να ήταν απλώς μια ένα τυχαίο γεγονό ότι συμπίπτει η υπογραφή του Βάτσλαβ Κλάου με τον εορτασμό των 20 χρόνων από την επανένωση της Ευρώπης. Πρέπει τώρα να πάρουμε τις αποφάσεις επί των προσώπων. Για τον πρόεδρο του Συμβουλίου και τον υψηλό τον είπα το εκπρόσωπο. Έχω να θέσω ένα ερώτημα σε εσά και να σα κάνω και μία αίτηση. Είσαστε έτοιμοι στι συζητήσει σα με του αρχηγού κρατών ε, και κυβερνήσεων να εξασφαλίσετε ότι υπάρχει μια κάποια ε, γεωγραφική ισορροπία που λαμβάνει υπόψη και τη Νέα Ευρώπη. Μήπως επίσης είστε έτοιμος να εξασφαλίσετε ότι θα υπάρχει μια μεγαλύτερη ε, παρουσία γυναικών στην Επιτροπή. Δεν φτάνει το ότι έχουμε την κυρία Βάστρομ. Ίσως θα πρέπει να υπάρχουν και περισσότερες γυναίκες σε υψηλό επίπεδο στην Κομισιόν. Δεν είναι για μένα κάτι το ορθό να έχουμε τόσες λίγες γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό δείχνει ότι δεν εκπροσωπούνται ισότιμα όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, εγώ δεν θεωρώ θα φταίτε εσείς αν δεν επιτευχθεί κάτι τέτοιο, αλλά θα ήθελα να σας ζητήσω πραγματικά να αγωνιστείτε για να υπάρχει μια καλύτερη γεωγραφική ισορροπία, μια καλύτερη ισορροπία των δύο φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε πράγματι να θεωρεί όλο ο πληθυσμός της Ευρώπης ότι εκπροσωπείται στην Κομισιόν. Επίσης, για τον ύπατο ε, εκπρόσωπο. Είπατε ότι θέλετε να προκρίνετε αυτή τη διαδικασία. Είσαστε σύμφωνος ότι θα πρέπει να υπάρξει πλήρης έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να αναλάβει τις εξουσίες του. Θα πρέπει λοιπόν ο υψηλός εκπρόσωπος, ο οποίος είναι και αντιπρόεδρο τη Κομισιόν και υπεύθυνο για τι εξωτερικέ υποθέσει Ευρωπαϊκή Ένωση να την χάνει, να απολαμβάνει τη υποστήριξη και τη έγκριση του Κοινοβουλίου. Εμεί σίγουρα θα διατηρήσουμε τι αρμοδιότητέ μα και θα υπερασπιστούμε τι εξουσίε μα, όπω είναι πολύ σαφέ, το κάναμε σαφέ στι συζητήσει μα με τον πρόεδρο τη Επιτροπή. Εμεί θα κρατήσουμε όλε αυτέ τι αρμοδιότητε άμομε, αλλά θέλουμε με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια δομή η οποία θα επιτρέψει να λειτουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο αναμένουν από εμά οι πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και μήνε. Το τελευταίο σημείο το οποίο θέλω να αναφέρω είναι το θέμα τη οικονομική και χρηματοοικονομική κρίση που ανέφερε ο κ. Ράιφερτ. Είναι κάτι το οποίο μα οδηγεί σε μεγάλε ανησυχίε. Πολύ σωστά τονίσατε ότι υπάρχει ο κίνδυνο να ανέβει ακόμα περισσότερο η ανεργία στην Ευρώπη. Εμείς λοιπόν δεν μπορούμε να άρουμε τα μέτρα υποστήριξης προς την οικονομία όσο δεν υπάρχει ανάκαμψη και στον τομέα τη ε, ανεργία. Γιατί αυτό περιμένουν και από εμά οι πολίτε να μην αποδεχτούμε σε αυτή τη νέα Ευρώπη να υπάρχει ένα τόσο ψηλό ποσοστό ανεργία. Επίση, υπάρχει το θέμα για την ενδεχόμενη φορολογία των χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Εδώ είναι απαραίτητο σε αυτή τη συζήτηση να τονίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι εμεί είμαστε έτοιμοι να ελέγξουμε τι ροέ κεφαλαίων, ότι είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα εργαλεία τα οποία θα μας βοηθήσουν και θα συμβάλλουν να χαλιναγωγηθεί η κερδοσκοπία στις χρηματαγορές και ότι δεν θα περιοριστούμε απλώς να βοηθήσουμε μία τράπεζα ή μία άλλη τράπεζα και με τον τρόπο αυτό να μην αποφύγουμε μελλοντικού μελλοντικούς στο μέλλον. Πιστεύω λοιπόν ότι ε, ένας τραπεζίτης ίσως θα πρέπει να κατανοήσει ότι δεν είναι μονάχα ένας ο οποίος δρά για τον δικό του λογαριασμό. Δεν είναι κάποιος ο οποίος μπορεί όπως έλεγε ένας παλιός τραπεζίτης να είναι ο τραπεζίτης στο όνομα του Θεού. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν και κάποια ευθύνη στο κοινωνικό σύνολο. Δεν είναι έργο του Θεού η χρηματοοικονομική δραστηριότητα. Είναι μια ανθρώπινη δραστηριότητα η οποία όμως θα πρέπει να συνοδεύεται με την προστασία από την κερδοσκοπία και την καταστροφή θέσεων απασχόληση και αυτό είναι απαραίτητο να γίνει στη σύγχρονη Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Σβόμποντα. Από τους ε, φιλελευθερούς τώρα, ο κύριος Γκίφερ Χοφστάτ. Πρόεδρε, αρχίζοντας θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Ράινφελντ και τη Σεσίλια φυσικά για την επικυρώση της συνθήκης της Λισαβόνας. Οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι έγινε χάρη στην αποφασιστικότητά σας, ε, χάρη στο πνεύμα, το συμβαστικό που σας διαπνεί. Υπήρχαν πολλοί ε, απεσιόδοξοι εδώ που πίστευαν ότι έπρεπε τελικά να περιμένουμε ε, τις εκλογές στη Μεγάλη Βρετανία και ότι δεν θα καταφέρναμε τελικά να επιτύχουμε την επικύρωση της συνθήκης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα κάνατε. Δέκα χρόνια εργασιών που εστέσαν με επιτυχία τελικά. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε επίσης και για τη σημερινή συζήτηση που δεχτήκατε να γίνει με τους αρχηγούς των πολιτικών ομάδων σχετικά με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον ΕΠΑΤΟ εκπρόσωπο και τη σύνθεση της νέας επιτροπής. Γιατί άλλη συζήτηση δεν πρόκειται να γίνει, δεν επικρατεί διαφάνεια. Ευτυχώς που υπάρχει ο τύπος για να μαθαίνουμε και τίποτα. Αλλά στο μέλλον ε, νομίζω πρέπει να το σκεφτούμε σοβαρά. Με ποιο τρόπο μπορούμε να φέρουμε ε, κάποια διαφάνεια σε μια διαδικασία που, α το παραδεχτούμε, είναι πάρα πολύ σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ακολουθήσω μια διαφορετική σειρά για να σχολιάσω τις διάφορες θέσεις. Εγώ θα αρχίσω με τη σύνθεση της Επιτροπής, Πρόεδρε, γιατί για το Κοινοβούλιο αυτό είναι το πιο σημαντικό ε, γιατί δική σας είναι η αρμοδιότητα, αλλά εμείς σας ελέγχουμε. Ε, ε, αυτό δεν συνισχύει με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Λοιπόν, τι σας ζητάμε συγκεκριμένα. Στην πρότασή σας ε, θα θέλαμε για πρώτη φορά να χρησιμοποιήσετε κλάστες ε, αγγλιστή, ομάδες για τις διάφορες αρμοδιότητες, δηλαδή να έχετε κάποιες θεματικές ενότητες ομαδοποίηση χαρτοφυλακίων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η εξωτερική δράση, η καινοτομία, ε, το ε, κλίμα και η αηφορία. Ε, κατά τα λοιπά, ε, οι οικονομικές υποθέσεις ε, και κατά τρίτον οι εσωτερικές υποθέσεις, δικαιοσύνη και τα λοιπά. Και γιατί να μην έχουμε αντιπροέδρους που θα ηγηθούν πραγματικά, θα επομιστούν την ευθύνη για αυτή την ομαδοποίηση των αρμοδιοτήτων που ε, είναι θέμα κοινή λογικής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έτσι θα βελτιώσουμε περαιτέρω την δράση της Επιτροπής υπό την Προεδρία σας. Δεύτερον, χρειαζόμαστε μια ισορροπία προς την αντιπροσώπηση των δύο φίλων στην Επιτροπή. Ε, και νομίζω ότι αυτό το θέμα σας απασχολεί και εσάς, ε, δηλαδή να έχουμε ε, και υποψήφιες για την Επιτροπή. Για τη θέση του υπάτου εκπροσώπου τώρα, κύριε Ράινφελ, το σημαντικό είναι να ε, γνωρίζουμε ποιο είναι ο στόχο. Συνεκτική πολιτική ΚΕΠΑ, συνεκτικέ κοινοτικέ πολιτικέ. Κάποιο που θα υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και σε κάθε δράση τη Ένωση ε, θα εισάγει αυτό το στοιχείο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και τρίτον, κάποιο ε, που θα υπηρετεί πραγματικά την εξωτερική δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά θα πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά αυτή τη προσωπικότητα ΚΕΠΑ, κοινοτικέ πολιτικέ, πολιτικές, ε, όλα αυτά θα πρέπει να ενωθούν, να ενοποιηθούν ε, ε, και θα είναι η αρμοδιότητα του Αντιπρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και η πιο σεξι σε εισαγωγικά υποψηφιότητα είναι αυτή του, για την θέση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Κύριε Ράινφελντ, ε, θα δώσω την άποψή μου. Έτσι μόνο άποψη μπορώ να δώσω για θα αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αλλά χαίρομαι που κάποιο από το Κοινοβούλιο θα μιλήσει ανοιχτά. Θέλουμε έναν ε, ε, προεδρεύοντα τη εργασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και όχι έναν πρόεδρο και θέλουμε κάποιον που πιστεύει στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ε, αν είναι να βγάλουμε πάπα, παίρνουμε ένα καθολικό. Εάν ε, τώρα αυτό που θέλουμε είναι πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ε, πρέπει τουλάχιστον να πιστεύει στην ιδέα της ευρωπαϊκής Ολοκλήρωση και όχι κάποιον ευρωσκεπτικιστή, γιατί ακούσαμε κάποια σχετικά πράγματα. Και τρίτον, για να είμαστε σίγουροι ότι πιστεύει στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, θα πρέπει να διαλέξουμε κάποιον που πιστεύει και στην κοινοτική μέθοδο εργασία, γιατί αυτή οδηγεί σε πρόοδο, όχι η διακρατική μέθοδο. Η διακρατική μέθοδο ε, είναι η ιδέα που χρησιμοποιούν κάποια κράτη και ευτυχώ κάποιε μεγάλε χώρε δεν πιστεύουν σε αυτό. Η διακρατική μέθοδο λοιπόν ε, του ευχαριστεί, αλλά όχι, Μιαζόμαστε κάποιον πιστεύει στην κοινοτική μέθοδο. Και τέλο, και θα κλείσω, ζητώ από τον κύριο Ράινφελντ να επιδιώξει μια συνενετική λύση προφανώς στο Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Συμμαχία που υπάρχει σε αυτό το κοινοβούλιο να αντανακλάται στους διορισμούς και στη σύνθεση. Ε, δηλαδή θέλουμε μια συμβαστική λύση ε, η οποία όμως θα αντανακλά αυτή την ε, φιλοευρωπαϊκή συμμαχία που θα οδηγεί σε πρόοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φερστάτ. Η κυρία Χάρμς, πρόεδρος της ομάδας των Πρασίνων, Ελεύθερη Ευρωπαϊκή Συμμαχία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Ράινφελτ, κύριε Μπαρόσο. Πιστεύω ότι είναι ακριβώς αυτή η ανάμνηση των ιστορικών γεγονότων που έλαβαν χώρα πριν από 20 χρόνια που τόνισε τη δυνατότητα να πραγματοποιηθούν οι πραγματικοί πόθη λαών που ίσως έπαιξε και κάποιο ε, ρόλο στην διαδικασία αυτή της ε, υπογραφής της ε, συνθήκης της Λισαβόνας από τον Βάτσλαβ Κλάους. Είδαμε τα λόγια, τα εμπνευσμένα του Βάτσλαβ Χάβελ που σίγουρα δεν μπορούν να συντεριαστούν με, μικρόψυχα παζαρέματα για άτομα και αξιώματα. Η διαδικασία αυτή λοιπόν της κύρωσης της συνδίκης Λισαβόνας χρειάστηκε 10 χρόνια, 10 χρόνια βασάνων και προβλημάτων που τελικά κατέληξαν στο να πιστούν όλοι οι ηγέτες κατών και κυβερνήσεων ότι αυτή είναι η σωστή οδός. Πρέπει να το ξέρουμε λοιπόν αυτό όταν ακούμε λοιπόν αυτά τα οποία ακούσαμε τον Βάτσλαβ Χάβελ και όταν τον έχουμε χειροκροτήσει όλοι σαν ενωμένοι ότι όλα αυτά τα πράγματα θα πρέπει να μας οδηγήσουν προς την κατεύθυνση που τόνισε. Αυτό που είναι απαραίτητο είναι να έχουμε μια ένωση, μια κοινή συμφωνία μεταξύ μας ότι είναι απαραίτητο στην κορυφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι στεναρά άτομα, στεναροί άνδρες και γυναίκες οι οποίοι θα οδηγήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι πραγματικά προς το συμφέρον των ε, ίδιων των κρατών που μπορεί να θέλουν μια πιο χαλαρή ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ δεν είμαι υπέρ μιας τέτοιας αντιμετώπισης Νομίζω ότι μέχρι στιγμής η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταφέρει να δείξει ότι είναι επιτυχής και αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω ότι αυτοί οι οποίοι παρουσιάζονται σαν υποψήφοι δεν είναι όλοι στο επίπεδο το οποίο για μένα θα ήταν απαραίτητο για να παίξουν αυτό το σημαντικό ρόλο. Επίσης και για το θέμα της Κοπενχάγης εγώ δεν μπορώ να συμμεριστώ τις απόψεις πολλών. Εγώ επανήλθα από την τελευταία συνδιάσκεψη προετοιμασία της Βαρκελόνης στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών και μέσα από την διάσκεψη αυτή έγινε φανερό ότι όλο και μικρότερες θα πρέπει να είναι οι προσδοκίες μας σε σχέση με τη διάσκεψη της Κοπενχάγης. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι λανθασμένο, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αποδεχθεί να πει ότι εμείς έχουμε κάνει όλα αυτά που περνούσαν από το χέρι μας και τώρα είναι απόκειται στους άλλους να κάνουν τα απαραίτητα. Αν εμείς λοιπόν δεν τηρήσουμε τις υποσχεώσεις μας για ένα πραγματικά αποτελεσματικό αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής, ποια είναι η ικανότητα πειθούς μας προς τους άλλους αν εμείς δεν εφαρμόσουμε αυτά τα οποία βρίσκονται στο δικό μας πακέτο. Ακόμα και αυτό το οποίο έχουμε συμφωνήσει δεν είναι επαρκέ για να τροχοπεδίσει την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη μας κάτω από τους 2 βαθμούς Κελσίου. Υπάρχει λοιπόν πραγματικά το ερώτημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε αν θέλουμε μια πραγματικά δεσμευτική νομικά ε, συμφωνία για τα θέματα αυτά ώστε να περατωθεί μια διαδικασία την οποία έχουν ζητήσει πάρα πολλοί Ευρωπαίοι στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δεν το κάνουμε αυτό λοιπόν πώς θα πάμε στην Κοπενχάγη και με τι προτάσεις θα μπορέσουμε να πούμε. Πάρα πολλές φορές λέμε ότι είναι απαραίτητο να έχουμε μια αηφόρο στρατηγική, μεγαλύτερη οικονομική και ενεργειακή αποτελεσματικότητα, πράσινη ανάπτυξη. Μια τέτοια λοιπόν νέα προσέγγιση στην Ευρώπη και ο Βάτσλαβ Χάβελ αυτό τόνισε και χειροκροτήθηκε για αυτό το στοιχείο. Αλλά η εντύπωσή μου είναι ότι αυτή τη στιγμή πολλές φορές οι Ευρωπαίοι μπορεί να το πράττουν φραστικά αυτό, να το υποστηρίζουν και να το χειροκροτούν δεν έχουν καταφέρει να το εφαρμόσουν σε πραγματικό επίπεδο και δεν έχουν κατανοήσει ακόμα ότι αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο θα μπορέσουν να δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης. Γιατί σίγουρα όταν έχουμε μια τέτοια οικονομική κρίση αυτό είναι ένας παραπάνω από χρόν λόγος να δώσουμε έμφαση στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Δεν είναι σαφές ότι η προσπάθειά μας για την ανάκαμψη είναι συγχρόνως και μια πορεία προς την αηφόρο ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ κύριε Χάρμς. Οι Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές, ο κ. Κέρκοπ έχει το λόγο. Θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ τη Σουηδική Προεδρία για τα βήματα προόδου ε, στον τομέα του κλίματος. Η αντιμετώπιση των κλιματολογικών αλλαγών είναι βασική προτεραιότητα και στον τομέα αυτό θα θέλαμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει κάθαρες και ε, σαφείς θέσεις. Το αποτέλεσμα μέχρι στιγμής δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πράγματι μπορεί να ε, ηγηθεί της προσπάθειας για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Τώρα έρχομαι στα θέματα του ΙΠΑ του εκπροσώπου για την εξωτερική πολιτική. Θα πρέπει να ορίσουμε πρώτα ακριβώς την φύση τη συγκεκριμένη αρμοδιότητα και μετά να αποφασίσουμε το πρόσωπο. Πριν πάρουμε μια τέτοια απόφαση, το Συμβούλιο στην ουσία προσκάλεσε να εκφραστεί ενδιαφέρον για υποψηφιότητες, όπου ίσως να εκφράστηκε και η υποψηφιότητα του κ. Φερχώστας. Ακούστηκαν προτάσεις από δεξιές αριστερέ κυβερνήσει, μικρές χώρες, μεγάλες χώρες, νότιες, βόρειες, αλλά κανένα δεν αναλαμβάνει την ευθύνη τελικά για το περιεχόμενο τη συγκεκριμένη αποστολή. Και μάλιστα και πολλοί προτείνουν η θέση αυτή να καταληφθεί ε, από πρόσωπα τα οποία προέρχονται μόνο από τη ζώνη ευρώ. Αυτό είναι μια σαφέστατη διάκριση. Εδώ τώρα γιορτάζουμε σήμερα μια μέρα 20 ε, χρόνια μετά από τα τραγικά γεγονότα που στήχησαν τόσο πολύ στην Ευρώπη. Γιορτάζουμε τα επιτεύγματα αυτών που καταπολέμησαν τον κομμουνισμό στην Πολωνία όπου ξεκίνησαν περίπου τα πάντα σε αυτή την κατεύθυνση την Ουγγαρία και στο τέλος και στο ίδιο το Βερολίνο. Είναι πάρα πολύ σωστό να πολεμά κανείς για την ελευθερία για όλους και όχι για ισχυρές θέσεις για ολίγους. Σας ευχαριστώ κύριε Κέκοπ. Ο κύριος Λόταρ Μπίσκι από την ομάδα της Νομόσπονδης Ευρωπαϊκής Αριστεράς, Πράσινης Φεδερικής Αριστεράς. Κύριε Πρόεδρε, έχει κυρωθεί η Συνδίκη Λισαβόνας και από τα 27 κράτη-μέλη. Ορισμένοι μπορεί να το γιορτάζουν αυτό σαν επιτυχία. Η δική μου ομάδα όχι. Έχω κατ' επανάληψη και κατά συρροή αναφέρει τους λόγους για το γεγονός αυτό και δεν θα το ξανακάνω τώρα. Ο λόγος είναι καταρχήν ότι η χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων έχει τύχει αυτοεξαίρεση τριών χωρών ήδη με οδηγίες σε αμφιβολίες. Και επίσης αν σκεφτούμε την ε, ομιλία του Βάτσλαβ Χάβελ και τον εορτασμό τον οποίο κάνουμε σήμερα για τα 20 χρόνια της κατάρρευσης του τείχους του Βερολίνου όλα αυτά μπορεί να φαίνονται ότι πράγματι είναι λόγος εορτασμού. Αλλά πιστεύω ότι πιο σημαντικό είναι να δώσουμε έμφαση στην ανάγκη να έχουμε μια πραγματική αηφόρο ανάπτυξη και ανάκαμψη από την κρίση. Το γεγονός ότι υπάρχουν περισσότερα δικαιώματα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τη συνθήκη της Λισαβόνα μπορεί να είναι θετικό. Αλλά από την άλλη πλευρά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα χρησιμοποιήσουν αυτή την ευκαιρία τη συνδίκησης τη Λισαβόνα για να ασκήσουν πιο συγκεκριμένε πολιτικέ και να αντιμετωπίσουν τα μεγάλα προβλήματα όπω είναι η κλιματική αλλαγή. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μια καλύτερη στρατηγική και να μπορέσει να παίξει ένα ηγετικό ρόλο, κάτι το οποίο δυστυχώ αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να συμβαίνει. Είναι απαραίτητο να τηρήσουμε την δέσμευσή μας, να μειώσουμε την ε, εκπομπή διοξιδίων του, διοξιδίου του άνθρακα και άλλων αερίων θερμοκηπίου είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν να αναλάβει και το βάρος των ευθυνών της για τη χρηματοδότηση των δράσεων προς την προστασία του κλίματος χωρίς να προσπαθήσει να βρει υπεκφυγές. Ο στόχος μας λοιπόν είναι όχι να αποφύγουμε η Σουηδία κάποια στιγμή να γίνει πάλι εινοπαραγωγός χώρα με την αύξηση της θερμοκρασίας. Είναι το θέμα να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την επιβίωση του ανθρωπίνου είδους και να αποφύγουμε καταστροφές, πλημμύρες και μετακίνηση τεράστιων ομάδων του πληθυσμού λόγω της κλιματικής αλλαγής. Όλα αυτά δεν είναι θέματα τα οποία μπορούν να επιληθούν σε εθνικό επίπεδο η προστασία του περιβάλλοντος, η καταπολέμηση της ένδυας και η ειρήνη είναι μεγάλες προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν δεν δράσει με ένα συνεκτικό τρόπο και υποδειγματικό στους τομείς αυτούς, δεν μπορεί κανείς να περιμένει να έχει η Ευρώπη <clears throat> να αποδοχεί σε διεθνές επίπεδο σε ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κόμις του μου θα έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, η νέα θέση του Πρόεδρου του Συμβουλίου με την οποία φαίνεται, στην οποία φαίνεται ότι όλοι εμένετε θα είναι ένας διορισμός για δύο χρόνια χωρίς καθορισμένες αρμοδιότητες. Οπότε θα πρέπει να λέτε στον κύριο Τόνι Μπλερ να μην στεναχωρηθεί πολύ άμα δεν πάρει τη θέση. Μετά από τη Λισαβόνα, ο πραγματικός Ρωμαίος αυτοκράτορας του 21ου αιώνα, ο Σάχης του 21ου αιώνα, θα είναι φυσικά ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο αγαπητός μας κύριος Μπαρόσο. Παρ' όλα αυτά, για το νέο ύπατο εκπρόσωπο, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Υπάρχει, θα έλεγα, ένα σαφής προϋπολογισμός, μεγάλος προϋπολογισμός για να δημιουργηθούν νέες ουσιαστικά πρεσβείες και αυτό είναι κάτι το οποίο απειλεί άλλωστε και τις θέσεις των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εσωτερικό του Συμβουλίου Ασφαλείας και αναφέραμε στη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία. Το πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι πάρα πολύ λίγες διπλωματικές αντιπροσωπείες αλλά πάρα πολύ άνεργοι. Γιορτάσαμε όλοι σήμερα τα 20 χρόνια από την πτώση του τείχους του Βερολίνου και καλά κάναμε. Αλλά τώρα έχουμε ένα νέο τείχος, όχι στα σύνορα, αλλά στο εσωτερικό των κρατών μας, στο εσωτερικό των χωρών μας και αυτό ακριβώς δεν το κατανοούν οι επαγγελματίες πολιτικοί του καθεστω, της τάξη. πολιτικής τάξης. Κύριε Βέρχοσταρτ έχουμε καθυστερήσει και γι' αυτό εμείς θα εξακολουθήσουμε για να μιλάμε στο όνομα του λαού της Ευρώπης και κατά των θεσμών που δεν πάβουν παρά να πλουτίζουν και θα συνεχίζουν να το κάνουν στο μέλλον και στερούνται φυσικά κάθε δημοκρατικής νομιμότητας. Ε, thank you. Σας ευχαριστούμε. Hans Peter Martin τώρα από τους, από τους Η δημοκρατία χρειάζεται επαναστάσεις. Αυτό πάντα ισχύει. Κύριε Δάρτμουθ, μιλήσατε για διαφάνεια και αναφερθήκατε και στον κύριο και ίσως θα μπορούσε και η Σουηδική Προεδρία να είναι ένα φωτεινό παράδειγμα. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν παίζει παιχνιδάκια για να θέτει άτομα τα οποία δεν είναι ικανά σε επίπεδο επιτρόπων και υψηλών εκπροσώπων. Η Γερμανία και η Αυστρία δίνουν αρνητικά παραδείγματα. Αλλά βλέπουμε εδώ στην ίδια αυτή την αίθουσα ικανά άτομα τα οποία δεν έχουν καμιά ελπίδα να φτάσουν στο επίπεδο των επιτρόπων. Γι' αυτό εμείς υποστηρίζουμε την ανάγκη να υπάρχουν σαφείς διαδικασίες για την επιλογή των επιτρόπων, διάφανος τρόπος και να υπάρχει πραγματικά η δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε τις ικανότητες και την γνώση που έχουν οι εκπρόσωποι των κρατών, οι εκπρόσωποι των λαών στον Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Πρωθυπουργό Φρέντερικ Ράινφελτ έχει το λόγο. Thank you very much for many, um, Σας ε, ευχαριστώ για τα αξιόλογα σχόλια και τις ενδιαφέρουσες ερωτήσεις που υποβάλλατε. Όπως είπε κάποιος, για να επικαιρώσουν τα, τη συνθήκη τα 27 κράτη-μέλη χρειάστηκαν πολλά χρόνια. Ε, και μετά ξαφνιάζομαι που μου με ρωτάνε τι θα γίνει μετά, εγώ δεν μπορώ παρά να βασιστώ στη συνθήκη για να εργαστώ. Το ε, σώμα φαστική σημασίας ε, φυσικά είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αυτό προβλέπεται ε, στη συνθήκη. Και πέραν τούτου είναι προφανές για μένα ότι είναι πρόβλημα πως διάφοροι υποψήφοι είναι οι πρωθυπουργοί κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και ε, αυτό είναι το πρόβλημα, δηλαδή θα περάσει κάποιος το μήνυμα ότι μπορεί να φύγει από τη χώρα του και μετά θα επιστρέψει και θα πει «Α, τελικά δεν θα φύγω». Είναι και αυτό ένας παράγοντας κάποια σημασία στην όλη διαδικασία. Για τον είπα το εκπρόσωπο, θα υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια, θα γίνει συζήτηση γιατί θα γίνουν ε, οι ακρόασεις ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριε Σφόμποντα, είναι σαφές ε, μέσα στη συνθήκη ότι ο ύπατος εκπρόσωπος αναλαμβάνει το αξίωμα ευθύς αμέσως αλλά πρέπει φυσικά να ανήκει στη νέα επιτροπή. Και όπως σας είπα και την προηγούμενη φορά εκεί είναι αυτονόητο, δεν το είχαμε προβλέψει να γίνει έτσι ακριβώς. Υποτίθεται ότι πριν αρχίσουμε τη Σουηδική Προεδρία έπρεπε να είχαν ρυθμιστεί αυτά τα ζητήματα. Τελικά, ε, πέραν κάθε προβλέψεως, ε, ήταν ιδιαίτερα χρονοβόρα η διαδικασία. Για το θέμα της ισορροπίας, γιατί είναι κάτι που ακούω επανειλημμένα, Σήμερα συγκεκριμένα έκανα ένα πρώτο γύρο διαπραγματεύσεων με τους 26 συναδέλφους μου. Ε, ε, μιλάμε για δύο θέσεις ε, και είναι δύσκολο να βρεθεί ισορροπία. Μιλήσατε για την γεωγραφική κατανομή, για τα φύλλα. Ξέρετε τι μου ζητάνε ως προς την ισορροπία ε, κέντρο-δεξιά και κέντρο-αριστερά. Ισορροπία ανάμεσα σε αυτά τα, στους δύο. Χρειαζόμαστε μεγάλη ισορροπία και πρέπει να συμμορφωθούμε με όλα τα κριτήρια που ε, αναφέρθηκαν είναι αυτονόητο ότι θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτύχουμε τη βέλτιστη δυνατή ισορροπία. θα μου ζητήσατε να κινηθούμε ταχύτατα και αυτό θα κάνουμε. αλλά ήθελα να σας πω ότι χρειάζεται χρόνος για τις ε, διαβουλεύσεις. Ε, δηλαδή, δύο ημέρες χρειάζομαι για να μιλήσω με τους υπόλοιπους 26 συναδέλφους μου. Είναι καταπληκτική ευκαιρία, αλλά χρειάζεται και χρόνος ε, για να τελεσφορήσουν οι διαπραγματεύσεις. Συμφωνώ με την ε, Ρεμπέκα Χάμσα ότι δεν κάνει αρκετά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε προβλέψει να ε, αυξήσουμε τις προσπάθειές μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να έχουμε νομικά δεσμευτικούς στόχους, αλλά χρειάζεται η αιρεσιμότητα. Και συμφωνούν οι συναδελφοί μου ως επιτοπλίστων. Ε, πολύ συγκεκριμένα λένε ότι για να καταφέρουμε περισσότερα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται να αναλυθεί αντίστοιχη δέσμευση και από τους λοιπούς εταίρους ανά τον κόσμο. Ε, οι αποφάσεις λαμβάνονται, ε, έχουμε πολλά παραδείγματα εθνικών ε, αποφάσεων. Στη Σουηδία παραδείγματος χάρη έχουμε ε, ως στόχο μέχρι το 2020 ε, μείωση 40%. Το ίδιο και στη Γερμανία πρέπει να καταφέρουμε περισσότερα πράγματα και δεν είμαι ε, εγώ αυτός που θα κατεβάσω τον πύχη στην Κοπενχάγη, αλλά ε, ε, πρέπει να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα για να κινηθούν και οι υπόλοιποι. Ε, πήγα στην Ινδία, στη ΣΥΠΑ, θα πάω στην Κίνα μέχρι το τέλος του μήνα. Χρειαζόμαστε συμφωνία για να λειτουργήσει ο μηχανισμός. Το δύσκολο είναι ότι η πρόκληση είναι παγκόσμιας κλίμακας, ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχα παγκόσμια ηγεσία ή παγκόσμια διαδικασία λήψης αποφάσεων όπως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και είναι δύσκολο να ληφθεί η απόφαση. Ξέρετε ότι ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το 13% των εκπομπών ε, και χρειαζόμαστε και άλλους για να τα καταφέρουμε. Χρειαζόμαστε τους υπόλοιπους εταίρους ε, και δεν μπορούμε να απόσχουμε από την ε, ε, συμφωνία, γιατί ποτέ δεν καταφέρουμε μόνοι μας να πετύχουμε αυτό το στόχο της, ε, του περιορισμού της αύξησης θερμοκρασίας σε λιγότερο από 2 βαθμούς Κελσίου. Τώρα γιατί χρειάζεται, μου είπατε, η καλύτερη εποπτεία των χρηματοπιστωτικών αγορών για να λειτουργούν πιο εύρυθμα οι αγορές θα αρχίσουν οι συζητήσει και θα συνεχιστούν υπό Ισπανική Προεδρία για το θέμα τη ανταγωνιστικότητα. Πώ μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα η αγορά εργασία, πού μπορούμε να εξέλθουμε από την κρίση τώρα που υπάρχουν τα πρώτα σημάδια τη ανάκαμψη. Σε μια ισορροπία χρειαζόμαστε ανάμεσα στα διδάγματα από το παρελθόν και για να λειτουργήσει η αισίωση για αγορά και την απόφαση που χρειαζόμαστε για να λειτουργήσει η καλύτερη αγορά της εργασίας και να έχουμε μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Πρωθυπουργέ. Τώρα καλώ στο βήμα τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Μπαρός. Πάρα πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε. Σχετικά τώρα με τις κλιματολογικές αλλαγές η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να καταλήξουμε σε μια δεσμευτική συνθήκη. Το, το ε, υποστηρίξαμε αυτό και στο Κιώτο, επικυρώσαμε το Κιώτο, τηρήσαμε το Κιώτο και είμαστε υπέρ μια δεσμευτική συμφωνία και για το μέλλον. Αν κάποιος δεν θέλει μια δεσμευτική συνθήκη, αυτός δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως η πραγματικότητα είναι ότι κάποιοι από τους πιο σημαντικούς μας εταίρους δεν είναι έτοιμοι ακόμα. Υπάρχουν δύο δυνατότητες δηλαδή. Από τη μία να παρετηθούμε λέγοντας ότι δεν θα πάνε καλά τα πράγματα ή από την άλλη να είμαστε ιδιαίτερα φιλόδοξοι για να πετύχουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα στην Κοπενχάγη. Και αυτό θα προσπαθήσουμε να επιδιώξουμε. Όσο πιο φιλόδοξοι μπορούμε να είμαστε θα το κάνουμε, θα είμαστε στην Κοπενχάγη. Αυτή είναι η στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτή είναι η στάση φυσικά της συνάντησης κορυφής αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων μια δεσμευτική συνθήκη η οποία να καθορίζει σαφώς τους στόχους και για τις αναπτυσσόμενες χώρες και σαφείς επίσης στόχους και για τις αναπτυγμένες χώρες που θα πρέπει να μοιράσουν τις ευθύνες οι οποίες υπάρχουν. Και θα πρέπει να υπάρξει χρηματοδότηση για τις φτωχότερες κυρίως υποανάπτυξη χώρες γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι χωρίς την υποστήριξη αυτή οι χώρες αυτές δεν θα είναι σε θέση να κάνουν τις προσπάθειες που απαιτούνται. Σχετικά με τα θέματα τα θεσμικά, εδώ θα ήθελα να είμαστε ε, σαφείς και ειλικρινείς. Είμαστε την παραμονή της θέσης σε ισχύ του νέου συστήματος. Ένα σύστημα ιδιαιτέρως απαιτητικό οι περισσότεροι από εμά κάναμε τεράστιες προσπάθειες για να έχουμε στη διάθεσή μας αυτή τη νέα συνθήκη. Τουλάχιστον για εννέα χρόνια μετά την οικία θέλαμε και ζητούσαμε μια πιο φιλόδοξη συνθήκη. Και τώρα πρέπει το νέο αυτό σύστημα να τεθεί σε ισχύ, να τεθεί σε λειτουργία. Είναι περίπλοκο γιατί η ένωσή μας είναι μια ένωση χωρών, μια ένωση κρατών, μια ένωση πολιτών Νομίζω ότι αυτό το οποίο έχει ε, σημασία εδώ είναι ο σεβασμός της συνθήκης. σήμερα μια κοινότητα δικαίου και την μέρα την οποία θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε με πλήρη ε, δεν θα μπορέσουμε μάλλον να λειτουργήσουμε με πλήρη σεβασμό της συνθήκης τότε θα έχουμε παραλείψει να φέρουμε εις πέρα στο καθήκον μας. Θα πρέπει λοιπόν να σεβαστούμε και τη συνθήκη και τις σαφείς αρμοδιότητες κάθε θεσμικού οργάνου, του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής κτλ. Εγώ είμαι ένας από αυτούς οι οποίοι θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προχωρά με ένα κυρίαρχο θεσμικό όργανο και μάλιστα με ένα θεσμικό όργανο το οποίο να εδρεώνεται εις βάρος των υπολείπων. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό. Αυτή η θεσμική ζήλια θα έλεγα είναι ίδιο των μετρίων. Νομίζω ότι αντίθετα εμείς θα ενισχυθούμε όλοι μαζί αν ενισχύσουμε ο ένας τον άλλον. Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε κάθε συμφέρον να έχουμε ένα ισχυρό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ισχυροποιείται μέσω της συνθήκης της Λισαβόνας ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με μια συνεκτική και ισχυρή ηγεσία και επίσης και μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία να είναι ισχυρή και σύμφωνη με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας, γιατί πολλά λέμε αλλά πολλά δεν διαβάζουμε μερικές φορές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φροντίζει και προστατεύει τα συμφέροντα της Ένωσης και είναι θεματοφύλακα της εφαρμογής της συνθήκης και των μέτρων που υιοθετούνται από τα όργανα της Ένωσης. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέει διαβάζοντας ο κύριος Μπαρόζο, πρέπει να επαληθεύει και να ελέγχει αν εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις της συνθήκης. Είναι αρμοδιότητες της συνθήκης αυτές οι οποίες αποδίδονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρέπει να τις ασκήσει. Αυτά όλα όμω θα πρέπει να γίνουν στα πλαίσια μια εταιρικότητα που να έχει σαν στόχο την ενίσχυση της Ευρωπαϊκή Ένωση, Εάν δεν έχουμε τα όργανα τα οποία να λειτουργούν σωστά, τι θα συμβεί. Τα κράτη-μέλη, ιδιαίτερα ορισμένα κράτη-μέλη, θα έχουν τάσει να λαμβάνουν αποφάσεις εκτός των οργάνων, εκτός της Ένωσης ίσως. Αυτό θέλουμε, όχι. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι οι αποφάσεις να λαμβάνονται στα πλαίσια τα θεσμικά, στα πλαίσια της κοινότητας δικαίου την οποία συναποτελούμε. Και αυτό θα ήθελα να σα πω και να ξεκαθαρίσω. Α ενισχυθούμε λοιπόν, α ενισχύσουμε ο ένας τον άλλον Ακούσαμε πραγματικά την εξαιρετική μαρτυρία του Βάτσλαβ Χάβελ σήμερα. Και όπως το έλεγε ο Ζωμονέ, τίποτα δεν γίνεται χωρίς τους ανθρώπους και τίποτα δεν διαρκεί χωρίς τους θεσμούς. Πρέπει λοιπόν τώρα να δημιουργηθούν ισχυροί θεσμοί, ισχυρά όργανα και αυτό θα το πετύχουμε μόνο στα πλαίσια του εταιρικού πνεύματος και γι' αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και για τις προτάσεις σας σχετικά με την οργάνωση και τη διάρθρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως και εσείς εγώ είμαι υπέρ της κοινοτική αντίληψης για τα πράγματα και υπέρ του σεβασμού της συνθήκης που κατανέμει σαφέστατα τις ευθύνε. Σύμφωνα με τη συνθήκη λοιπόν ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία της και φυσικά θα αναλάβω τις ευθύνε μου. Όταν παρουσιάσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σαν ένας απλός χειροτέχνης αν θέλετε, θα προσπαθήσω να ευχαριστήσω μεν αυτούς που με βοήθησαν, αποδεχόμενος όμως για το τελικό προϊόν της προσπάθειάς μου τη πλήρη ευθύνη. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι να το κατανοήσουμε όλοι ότι ο καθένας θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του και αυτό θα πρέπει να το κάνει στα πλαίσια του σεβασμού των υπολείπων οργάνων και έχοντας σε ανώτατο επίπεδο φυσικά το ευρωπαϊκό συμφέρον. Ευχαριστώ Πρόεδρε για την παρουσίασή σας και τις παρατήρησεις σας. Τώρα θα περάσω στους υπόλοιπους ομιλητές και θα ξεκινήσω με τον Ίνιγκο Μέντες Δεβίγκο δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι συγχαίρει τον κύριο Ράινφελτ γιατί έφερε σε ασφαλή λιμένα το πλοίο της Λισαβόνας. είναι σαν μια ιστορία σαν τον γέρο και τη θάλασσα του Χέμιγουε που τελικά γυρίζει η βάρκα στο λιμάνι της. Λοιπόν δεν έφτασε πραγματικά η συνθήκη της Λισαβόνας τόσο εύκολα στο λιμάνι, αλλά διέσωσε ο ψαράς τουλάχιστον το σκελετό της. Νομίζω ότι από όλους υπήρξε ένα πνεύμα επίτευξη συμβιβαστικών λύσεων με τον πρόεδρο της Τσεχικής Δημοκρατίας. Μας ενόχλησε μας το κοινοβούλιο αυτό το οποίο έγινε, αλλά σε τελική ανάλυση, όπως λέει και η Ισπανική παροιμία, τέλος καλά, όλα καλά. Υπάρχει τώρα η συνθήκη η οποία είναι σε εφαρμογή και πρέπει να σκεφτούμε για το πώς θα την εφαρμόσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Εγώ δεν θέλω να δώσω συμβουλέ στον κύριο Μπαρόσο για το πώ θα συνθέσει την Επιτροπή του. Σέβομαι την αυτονομία και την ανεξαρτησία του Προέδρου της ε, Κομισιόν που έχει την ικανότητα να πράξει όλα αυτά τα οποία είναι απαραίτητα. Είναι δική του ευθύνη να παρουσιάσει το σώμα των Επιτρόπων και εμεί θα πρέπει όταν παρουσιάσει την Επιτροπή να κρίνουμε υπέρ ή κατά. Ούτε έχω να δώσω και συμβουλέ στον Πρόεδρο του Συμβουλίου. Απλώ θέλω να του υπενθυμίσω κάτι το οποίο έγινε κατά τη διάρκεια των ε, εργασιών της ε, συνταγματικής συνέλευσης. Στο πρώτο σχέδιο που αναφέραμε ότι πρέπει να υπάρχει ένας πρόεδρος του Συμβουλίου, η πρότασή μας ήταν ο πρόεδρος του Συμβουλίου να είναι ένας πρωθυπουργό, ο οποίος να έχει ασκήσει το αξίωμα αυτό τουλάχιστον 2,5 χρόνια. Ήταν η λεγόμενη ρήτρα Τζον Μπρούτον, όπως την λέγαμε εμείς γιατί έτσι τότε θα μπορούσε ο Τζον Μπρούτον που είχε μείνει στην εξουσία δύο χρόνια και εφτά μήνες να είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά σήμερα αναρωτιόμαστε τι σημαίνει το να είναι κανείς πρωθυπουργό. Γιατί έχει κάτι περισσότερο από τους κοινού θνητούς. Γιατί πρέπει ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Συμβουλίου να είναι ένας πρώην πρωθυπουργό. Κύριε Ράινφελτ, μήπως είναι καλύτερο να βρείτε ένα άτομο το οποίο είναι το καλύτερο άτομο για να εκπροσωπεί το ηθικό ανάστημα και τις, τα επιτεύγματα της ε, Ευρώπης. Έχετε και ένα όπλο στη διάθεσή σας που είναι ότι η εκλογή του Προέδρου του Συμβουλίου δεν είναι υποχρεωτικό να γίνει με ομοφωνία αλλά με ειδική πλειοψηφία. Ή δυνατόν λοιπόν συνένεση, εάν όχι όμως χρησιμοποιήστε το όπλο της ειδική πλειοψηφίας για να βρείτε τον καλύτερο δυνατό Πρόεδρο του Συμβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Μέντας Ντεβίγο. Το λόγο έχει η κυρία Ουλτσβοκ για 1,5 λεπτό. Πρόεδρε, χαίρομαι πάρα πολύ που ε, εξεδήλωσε η Σουηδική Προεδρία τη φιλοδοξία της ε, να επισπεύσει τις προσπάθειες ε, για τη στρατηγική εξόδου ε, ούτως ώστε να μην να μην παγιωθεί η υψηλή ανεργία στην Ευρώπη. Με ανησυχία ότι όλοι μας προειδοποιούν ότι η σύνοδος της Κοπενχάγης δεν θα στεφτευτεί με επιτυχία τελικά και θα ήθελα να το σχολιάσει περαιτέρω ο κύριος Ράινφελντ. Ε, αυτό φαίνεται και στα συμπερασμάτα του τελευταίου Συμβουλίου. Ε, ο, οι αναπτυγμένες χώρες πρέπει μέχρι το 2005 να μειώσουν τις εκπομπές κατά 80 με 95% κανονικά. Αλλά καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά χρειάζονται ισχυρή δέσμευση. Ε, και επίσης υπάρχει το θέμα της χρηματοδότησης ε, των προσπαθειών που θα κάνουν οι αναπτυσσόμενες χώρες γιατί εκείνες έχουν συνεισφέρει και ελάχιστα σε σχέση με εμάς ε, στις κλιματικές αλλαγές και πρέπει να κάνουν τώρα τις σοβαρέτερες προσπάθειες και δεν καταφέρνουν να συμφωνήσουν στο Συμβούλιο για τη χρηματοδότηση. Η η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποσχεθεί, όπως μας είπε ο, ο κύριος Ράινφελτ, να κάνει την δέουσα ε, συνεισφορά για την καταπολέμηση των ε, κλιματικών ε, αλλαγών. Αλλά συγγνώμη, αυτό είναι παράλογο. Ε, δηλαδή θα πρέπει να κάνει μια σοβαρή προσπάθεια και όχι αυτά που μας προτείνει ο κύριος Ράινφελτ. Μας είπε ο κύριος Ράινφελτ ότι θα ε, δαπανηθούν 57 δις ε, τα πρώτα χρόνια. Συγγνώμη, αλλά αξίζει έστω και να αναλυθεί μια τέτοια δέσμευση. Δεν λύνει το πρόβλημα. Και τι, τι κάνουμε με τα προβλήματα που έχουμε με τη ΣΥΠΑ, με την Κίνα, με την Ινδία έχουν εξαιρετικό πρόβλημα με την άκαμπτη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό και ε, αν είχε δεήσει να παραμείνει εδώ στην αίθουσα ο κύριος Δράινφιλ θα μπορούσα να του θέσω πάρα πολλές τέτοιες ερωτήσεις ε, γιατί μιλάμε για μεγάλη πρόκληση ε, η Σύνοδος της Κοπενχάγης και δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε να αποτύχει. Ευχαριστούμε κυρία Ούλφσκογκ. Ξεπεράστε το χρόνο σας, αλλά θα προλάβουμε την επόμενη φορά ίσως. Δίνω προηγουμένως το λόγο στον κύριο Λάμπς για ένα λεπτό. Χαιρόμαστε όλοι για το γεγονός ότι έχει κυρωθεί η συνθήκη της Λισαβόνας. Όλο αυτό θα πρέπει να είναι μια ευκαιρία για περισσότερη δημοκρατία, περισσότερο έλεγχο και στον υψηλό εκπρόσωπο. Ο πρόεδρος όμως του Συμβουλίου θα πρέπει να ξέρει ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει και έλεγχος από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Θα πρέπει να είναι ένας πραγματικός διαμεσολαβητής των, ε, μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό το οποίο είναι απαραίτητο καταρχήν για να πετύχει κάτι τέτοιο να υπάρχει συνένεση του Συμβουλίου. Όταν θέλουμε να εκλέξουμε ένα Πάπα πρέπει να είναι καθολικό. Όταν θέλουμε να εκλέξουμε ένα πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα πρέπει να έχουμε κάποιον ο οποίο έχει ευρωπαϊστικό πνεύμα και πιστεύει πράγματι στην προσέγγιση τη Ευρώπη. Πρέπει και πάλι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να φέρεται ευρωπαϊκά, ευρωπαϊστικά. Αυτή η συζήτηση η οποία γίνεται σήμερα δεν θα είχε γίνει αν δεν την είχε ζητήσει η φιλελεύθερη ομάδα. Θα γινόταν μόναχα στα μέσα ενημέρωση, ίσω στους ε, διαδρόμους. Κύριε Ράινφελ, δεν είναι μονάχα ένα θέμα ισορροπίας μεταξύ κέντρου αριστεράς και κέντρου δεξιάς, είναι μια ισορροπία μεταξύ κέντρου αριστεράς και δεξιάς. Ευχαριστώ συνάδελφε. Δίνω το λόγο τώρα για Νίκ Ζαντότ. 300.000 νεκροί λόγω των κλιματολογικών αλλαγών. Η αδράνεια είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Ξέρουμε ποια είναι τα προβλήματα, παρόλα αυτά οι διαπραγματεύσεις δεν προχωρούν. Είναι εύκολο να λέμε φυσικά ότι φταίνε οι Ηνωμένε Πολιτείε. Παρόλα αυτά εμείς θεωρούμε ότι η ευθύνη της Ευρώπης είναι τεράστια. Η Ευρώπη δεν είναι πια αντίθετα από αυτά που έλεγε ο Προεδρεύων, ο ηγέτης στον τομέα της διαπραγμάτευσης για τις κλιματολογικές αλλαγές μέχρι το τέλος του αιώνα θα υπάρξει αύξηση της μέσης θερμοκρασίας λόγω των κλιματολογικών αλλαγών κατά 4 βαθμούς. Αυτό είναι απαράδεκτο και δεν θα πρέπει να κρυφόμαστε πίσω από τον αυστηρά νομοθετικό χαρακτήρα αυτής της απόφασης. Ανεξάρτητες μελέτες δείχνουν σήμερα ότι η Ελβετία, η Νορβηγία, η Ιαπωνία κάνουν προσπάθειες ανώτερες της Ευρώπης. Από τις αναδυόμενες χώρες η Βραζιλία, η Ινδονησία η Ινδία αναλαμβάνουν ε, δεσμεύσει σε εσωτερικό επίπεδο υψηλότερε από αυτέ τι οποίε συζητά η διεθνή επιστημονική κοινότητα. Από αυτά που είπε ο Βάσλατ Χάβελ, αυτό το οποίο βγάζουμε είναι ότι πρέπει να είμαστε μετριόφρονες και ρεαλιστέ. Α μην λέμε ότι μόνο στην Ευρώπη τα πράγματα πηγαίνουν καλά, ότι τίποτα δεν άλλαξε από το Κιώτο κτλ. Και, και η Ευρώπη είναι πάντα πρόδρομο. Όχι. Εμείς αρνούμεθα να λάβουμε υπόψη μας τις απόψεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και φταίει το Συμβούλιο γι' αυτό ανέλαβε την ευθύνη της αποτυχίας της Κοπενχάγης. Παρ' όλα αυτά υπάρχει χρόνος. Μπορεί να ανακτήσει την ηγέτιδα θέση της η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκοντας ακριβώς με 30 δις τις χώρες του Νότου. Αυτό θα οδηγήσει σε μια συμφωνία και με τους Αμερικανούς. Ευχαριστώ κύριε Ζαντό. Για ένα λεπτό τον λόγο στον κόνομα Τσιμάνσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα συμπεράσματα της, ε, του Συμβουλίου του μηνός Οκτωβρίου είναι μια καλή ευκαιρία για να επανεξετάσουμε τη θέση μας στα πλαίσια των κλιματολογικών αλλαγών οι συνέπειες μας θα πρέπει φυσικά, οι συνέπειες μάλλον των δράσεών μας συνδυάζονται με τις αντίστοιχες συνέπειες των αποφάσεων και των δράσεων των Κινέζων και των Αμερικανών και άλλων χωρών. Δεν θα πρέπει εμείς να καταστρέψουμε την οικονομία μας αντίθετα από αυτά τα οποία θα κάνουν άλλες χώρες. Αν υπήρχε οικονομική ανάπτυξη αυτή την εποχή θα ήταν πιο εύκολη η προσπάθεια. δεν θα πρέπει να δημιουργηθεί μια κατάσταση όπου κάποια κράτη-μέλη θα πληρώνουν διπλά στα πλαίσια του συστήματος ανταλλαγών εκπομπών και από την άλλη να πληρώνουν και για την επιδότηση άλλων χωρών. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Ο κύριος Μποργέζιο, δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εδώ και λίγες μέρες μια πολύ σοβαρή απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του Στροσφούργου σημείωσε και υπογράμμισε μια κατάσταση πάρα πολύ σοβαρή. Γύρω από την κατάσταση αυτή έχει εκφραστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ιδιαίτερα επιφυλακτικά. Και αναφέρομαι στην απόσυρση των σταυρών από τις σχολικές τάξεις στα δημόσια σχολεία της Ιταλίας. Πρόκειται για μια σαφέστατη παραβίαση και της αρχής της επικουρικότητας. Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, λέει ο κύριος Μποργέζιο. Και θα πρέπει να δούμε τι συνέχεια θα δοθεί στην υπόθεση αυτή με την υιοθέτηση της συνθήκης της Λισαβόνας. Ελπίζω να μην συνεχίσουμε σε αυτήν την απαράδεκτη λογική ενός ευρωπαϊκού δικαίου που καταπνίγει και στρεβλώνει τις ευρωπαϊκές ένομες τάξεις των μεμονωμένων χωρών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έπρεπε να αντιδράσει με πολύ πιο σκληρό τρόπο γιατί μία απλή προφορική θα έλεγα καταγγελία δεν αρκεί. Οι περισσότερες από τις Ιταλικές πολιτικές δυνάμεις που εκπροσωπούν την ευαισθησία του λαού μας εκφράστηκε και νομίζω ότι το θέμα δεν είναι μόνο πολιτικό, είναι και πολιτιστικό όπως έλεγε ένας μεγάλος φιλόσοφος ο οποίος έλεγε ότι υπάρχουμε και υπάρχουμε και είμαστε χριστιανοί. Εν πάση περιπτώσει Ακούγονται πάρα πολλές απόψεις, γίνονται πάρα πολλές ε, συναντήσεις για λόγους ιστορικούς. Ε, διαρωτώ όμως, βλέποντας τα ονόματα τα οποία κυκλοφορούν, Μπαλκενέντε, Μίλιμπαντ και Βαν Ρόμπουι. Κανένας δεν έχει παρατηρήσει μέχρι τώρα ότι και οι τρεις ε, αυτοί συχνάζουν στη σχέση, στη λέσχη μάλλον Πίλτεμπεργκ ή στην τριμερή συνάντηση. Καταλαβαίνετε ότι εδώ πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια, να μάθουμε περισσότερα πράγματα και θα πρέπει να ζητήσουμε από τα συγκεκριμένα αυτά πρόσωπα αν είναι υποψήφοι των χωρών τους, των πολιτικών τους δυνάμεων ή αυτών πραγματικά των μυστικών υπηρεσιών και ομάδων που αποφασίζουν και συνομωτούν πίσω από τους πολίτες της Ευρώπης. Ευχαριστώ κύριε Μπορκέζιο. Ο Σώσα Βάγνερ. Ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, μπορέσαμε να ξεπεράσουμε την γενική αβεβαιότητα και ανησυχία με την έγκριση και την κύρωση της συνθήκης της Λισαβόνας. Τώρα είναι ο καιρός να σκεφτούμε ποια θα είναι η αντιμετώπιση που θα υπάρχει στο μέλλον για τις εθνικιστικές δράσεις που τόσο πολύ εμποδίζουν την ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Πιστεύω ότι αυτές οι μορφές κλειδονισμών δεν μπορούν να συνεχίσουν ατιμωρητοί. Είναι απαραίτητο με ψυχραιμία να σκεφτούμε τι μέτρα θα μπορέσουμε να αναλάβουμε για τα επόμενα χρόνια για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις κινήσεις. Θέλουμε να έχουμε ένα πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ο οποίος θα είναι ένας άντρας ή ακόμα καλύτερο μια γυναίκα πεπισμένη για την ανάγκη του Ευρωπαϊκού Φεδεραλισμού που υποστηρίζει το ευρώ που είναι μέσα στο χώρο του Σέγγεν και που ταυτίζεται και δεσμεύεται με την Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε. Θα ήθελα να σας πληροφορήσω συναδέλφοι ότι μια αντιπροσωπεία της Μαλαισιανής Ομοσπονδίας είναι παρούσα στα επίσημα θεωρία. Θα ήθελα να ευχηθώ το καλωσόρισε σε αυτήν την αντιπροσωπεία που καθοδηγείται από τον πρόεδρο της Γερουσίας της Μαλαισίας Φον Μέγκ. Οι σχέσεις ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κοινοβούλια της Μαλαισίας είναι τακτικές. Είναι μια ζωηρή κοινωνία η Μαλαισία, μια ζωηρή οικονομία επίσης και ιδιαίτερα δραστήρια στα πλαίσια του ΑΣΕΑΝ. Γι' αυτό ακριβώς είναι μεγάλη χαρά που καλωσορίζουμε τους μαλαισινούς φίλους. Ελπίζουμε η επίσκεψή σας να είναι καρποφόρα και ενδιαφέρουσα. Δίνω τώρα το λόγο στον κύριο Μπροκ για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε,